good afternoon everybody. Let's start our... Καλησπέρα σε όλου. Ε, άρχεται η την μα συνεδρίαση. Καταρχήν θα ήθελα να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη θεσινή συνεδρίαση. Υπάρχουν αντιρρήσει. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Έλαβα αίτημα της ΑΛΤΕ για διορισμό του κυρίου Κέντ Γιώχανσον ως μέλος της διακοινοβουλευτική αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κροατία.